Κόζα. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ τον Επίτροπο Μίμητσα να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Περίπου αυτή την εποχή πέρσι υπήρξε η τελευταία χώρα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κύρωσε την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι προσελεωμένα στο εξή μήνυμα. Δεν θέλουμε να προσαρμόσουμε τους ανθρώπους στο περιβάλλον τους. Αντιθέτως, θέλουμε να προσαρμόσουμε το περιβάλλον στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Και αυτό το ακριβώς θα κάνει και η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσβασιμότητα. Έπειτα από τρία σκληρά χρόνια διαπραγματεύσεων, έπειτα από ένα σκληρό παζάρι, καταφέρατε να καταλήξετε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το πολύ σημαντικό ε, ε σε αυτή τη πολύ σημαντική νομική πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λόκιγκαρ, τον κύριο Κόσα, τον κύριο Τέιλορ για το γεγονός ότι αυτό που έχουμε πλέον επιτάπητος είναι ένα ισχυρό πακέτο που θα καταστήσει την Ευρώπη πιο προσβάσιμη για ζωή αλλά και για εργασία για τα άτομα με αναπηρίες. Η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία της Κομισιόν στον κοινωνικό τομέα. Το Σεπτέμβριο του 2017 είχαμε υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση η οποία περιλάμβανε ομοιόμορφη εφαρμογή και κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριλάμβαναν ε, τους αντίστοιχους κανόνες της σύμβασης του ΟΗΕ που βασίζονταν στις, ε, στα ισχυρά σημεία της ενιαίας αγοράς μας. Με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για προσβάσιμες ε, υπηρεσίες και προϊόντα. Ο ίση όροι ανταγωνισμού που δημιουργήσαμε είναι ωφέλιμη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί αυτό θα καταστήσει τα τα προσβάσιμα προϊόντα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες πιο οικονομικά προσιτές. Αυτό θα επιτρέψει σε πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων, να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασίας, επί ίσης όρης με όλους τους συμπολίτε τους. Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα θα καλύπτει ε, μια τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, τερματικά πληρωμών, τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Πρόσβαση σε οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικό εμπόριο, κάποιες υπηρεσίες μεταφορές, μεταφορών. Αυτές είναι σημαντικές υπηρεσίες και σημαντικά προϊόντα για την καθημερινότητα των πολιτών, που όλο ένα και περισσότερο ε, επηρεάζονται από την ψηφιοποίηση. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η πράξη προσβασιμότητας θα συμβάλλει και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την ε, πρόβλεψή του για, την, για τον μη αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. Θέλουμε επίσης οι κανόνες να είναι μελλοντοστραφείς, ανθεκτικοί στο μέλλον, και να εξασφαλίσουμε ότι η ψηφιακή επανάσταση θα αποτελέσει καταλήτη υπέρ της ε, κοινωνικής ένταξης και ότι δεν θα μείνει κανείς απ' έξω. Θα πρέπει όλα αυτά βεβαίως να ειδωθούν υπό το πρίσμα και άλλων ευρωπαϊκών μηχανισμών όπως ή νομικών πράξεων, όπως είναι η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες ή η οδηγία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες όπου η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση η πράξη για την προσβασιμότητα θα βοηθήσει στην εφαρμογή όλων αυτών. Θέλω τέλος να τελειώσω ότι ο αντίκτυπος αυτής της πράξης υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της. Οι απαιτήσει που περιλαμβάνει για την προσβασιμότητα μπορούν να εμπνεύσουν και άλλους κλάδους και άλλες περιφέρειες του πλανήτη. Στόχος της Ευρώπης είναι να γκρεμιστούν τα σύνορα μεταξύ χωρών και λαών. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία για να κατεδαφίσουμε τα εμπόδια που περιόριζαν τα άτομα με ανεπηρία όσον αφορά τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή και στην αγορά εργασία. Σας ευχαριστώ και βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη υπέρ αυτής της πράξης προσβασιμότητας που θα επιφέρει σημαντικότατε θετικέ αλλαγές στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Ευχαριστώ τον Επίτροπο κ. Μιμίτσα για την Επιτροπή Πολιτισμού. Η κυρία Βόρντ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύριο άνθρωποι με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας αριθμός που αναμένεται να φτάσει 120 εκατομμύρια μέχρι το 2020. Άνθρωποι με αναπηρίες στην Ευρώπη πολύ συχνά έχουν πρόβλημα να έχουν πρόσβαση σε πολύ βασικά προϊόντα και υπηρεσίες επισοτήμου βάσεως με τους άλλους. Ε, αυτό σημαίνει καθημερινό αποκλεισμό από την κοινωνία και από τη χρήση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών κάτι το οποίο θεωρείται σαν δεδομένο από την πλειοψηφία. Όπω να πάει κανεί στην τράπεζα, να αποσύρει χρήματα από ένα αυτόματο μηχάνημα, να μπει κανεί σε πανεπιστήμιο, σχολείο, σε βιβλιοθήκη, σε θέατρο ή οδήποτε δημόσιο κτίριο, χρήση του υπογείου, η αγορά ενό εισιτηρίου. πρεπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, με περισσότερε επαφέ με τι κοινωνίε των ανθρώπων με αναπηρία, να ακούσουμε τι ανάγκε και να δράσουμε βάσει των καθημερινών του εμπειριών. Κανεί να μείνει έξω, κανείς να μείνει πίσω σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Περί αυτού πρόκειται αυτή η έκθεση. Τίποτα γύρω από μας χωρίς εμάς, όπως λένε οι άνθρωποι με αναπηρία, οι φίλοι μου. Και θα θέλουν να έχουμε καλά αποτελέσματα όταν θα ψηφίσουμε την έκθεση και δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Τζούλη. Τώρα Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητα των Φίλων. Στάσφερκουτ, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Α, δεν είναι εδώ. Επόμενος ο μιλητής. Που θα αναφερθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Έχει το λόγο για ένα λεπτό, κυρία Κούνεβα. Το πρόεδρε έξι χρόνια πέρασαν από την αναγγελία της επιτροπής για την ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. σήμερα καλούμαστε να την ψηφίσουμε πιο αποδυναμωμένη από ποτέ γιατί δεν ακούστηκαν οι φωνές των ατόμων με αναπηρία. προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε τις προτάσεις του αναπηρικού κινήματος μέσα από εκατοντάδες τροπολογίες αλλά οι συντηρητικές δυνάμεις του κοινοβουλίου τις καταψήφισαν. έτσι δεν έχουμε προσβάσιμο δομημένο περιβάλλον ούτε διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. το χειρότερο χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα έξι χρόνια μέχρι να δούμε την οδηγία να εφαρμόζεται. τι προσβολή για το αναπηρικό κίνημα είναι αυτό! όμως εμείς σεβόμαστε τους φορείς αναπηρίας. γι' αυτό και θα συνεχίσουμε τον αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ μέχρι να άρουμε όλα τα εμπόδια. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες για το ΕΛΚ. Συνάδελφε Σβάμπ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι και εγώ που τα καταφέραμε να ανταποκριθούμε στο καθήκον θέσπισης κανόνων για την άρση των εμποδίων, για την προσβασιμότητα, γιατί όπως υπόθηκε 80 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προβλήματα κινητικότητας, αναπηρίες στην Ευρώπη, γι' αυτό και οι, άνθρωποι, αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό ε, απαιτεί να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους τους φορείς λειτουργίας ε, υποδομών και θεωρώ ότι με αυτό που κάναμε σήμερα έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτόν τον στόχο. Και ε, θεωρώ ότι ταυτόχρονα με την κοινωνική διάσταση δημιουργούμε και πολύ σημαντική βασικά οικονομικά κριτήρια. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εξαιρούνται από τους κανόνες αυτούς οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί θα ήταν δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο και θεωρώ ε, επίσης ότι το δομημένο περιβάλλον το οποίο ήθελε να ζητήσει το που ζητούσε το κοινοβούλιο να συμπεριλαμβάνεται δεν έγινε κατόρθωτο κάτι τέτοιο αλλά δεν πειράζει την επόμενη φορά. Ξανέλαβα δύο λεπτά παρακαλώ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και σε προϊόντα είναι κάτι φυσιολογικό για το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, αλλά μπορεί να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τα 4 εκατομμύρια αναπήρους που έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές ελπίδες από το κείμενο αυτό. Η πράξη όμως για προσβασιμότητα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Χρειάστηκαν πρώτα απ' όλα 10 χρόνια για να παρουσιαστεί η πρόταση και 4 χρόνια για διαπραγματεύσει. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε στα μέσα του δρόμου ακόμα. Μόνο μερικέ είναι οι επιτυχίε και ευχαριστώ του συναδέλφου, κυρίω στον ψηφιακό τομέα. Η πράξη θα έπρεπε να φροντίσει περισσότερο για την πρόσβαση με τερματικά πληρωμών ε, μέσω υπολογιστών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και πλήρης κινητικότητα, να μπορεί δηλαδή πλήρως ο ανάπηρος να ταξιδέψει παντού, να φτάσει στα μαγαζιά. Η πράξη αυτή προσβασιμότητας δεν βρίσκεται στο ύψος των προστοκιών μας. Πολλές φορές επικρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αποφάσεις που είναι εκτός πραγματικότητας. Οι χώρες μέλη είναι αυτές που πήραν την απόφαση να μειώσουν το κόστος και να αγνοήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει προηγουμένως για την προσβασιμότητα. Για μας, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η χρήση προϊόντων και υπηρεσιών από όλου τους πολίτες εξίσου είναι κάτι θεμελιώδες. Εμείς πιστεύουμε ότι αποτελεί μία προϋπόθεση συνεκβάνου για την ενσωμάτωσή τους, την ένταξή τους στην κοινωνία. Οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, όλοι αυτοί που δυσκολεύονται. Συνεπώς δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. Ευχαριστώ για τους συντηρητικού. Συνάδελφε Σιτνάσκα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι η οδηγία αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ θετική συμβάλλει στη βελτίωση της, ε, των όρων ζωής και εργασίας ε, των ατόμων με αναπηρία. Και για το γεγονός βεβαίως ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα εντός της θητείας. Από την αρχή είχα εκφράσει την πλήρη υποστήριξή μου στην πρόταση οδηγίας αυτή της Κομισιόν και σε συνεργασία με τους συναδέλφους προσπάθησα να βελτιώσω το κείμενο. Οι δε διαπραγματεύσει που ακολούθησαν την υποβολή τη πρόταση από την Κομισιόν θεωρώ ότι άλλαξαν το περιεχόμενο τη οδηγία και δυστυχώ τελικά καταλήξαμε με ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν τόσο φιλόδοξο, όχι μόνο τόσο φιλόδοξο όσο θα ήθελα εγώ, αλλά όσο κυρίω οι επιθυμίε ε, των, ε, όσο επιθυμούσαν οι άνθρωποι με αναπηρίες. Βεβαίως δεν είμαστε στο τέλος του δρόμου. Σήμερα δεν χρειάζεται να είμαστε απεσιόδοξοι. Νομίζω ότι το ζήτημα της προσβασιμότητας θα συνεχίσει να μας απασχολεί και τα επόμενα χρόνια, ιδίως στο πλαίσιο των κρατών μελών. Ο κύριος Σόλτες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως υπόθηκε, πάνω από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ε, ζητούν και περιμένουν αυτήν την ε, νομική πράξη να θεσπιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική του δουλειά. Καταρχάς, την, την, η, η πράξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως ε, πρόκειται, όπως υπόθηκε, μόλις για το πρώτο βήμα. Δεν καλύπτει, ούτε ανταποκρίνεται, ούτε ικανοποιεί η οδηγία αυτή όλα τα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί. Όμως βρισκόμαστε σε ένα σημείο εκκίνησης. Είναι μια αφετηρία και νομίζω ότι με ελπίδα μπορούμε να αποδείξουμε και να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους ακούει. Κούσαμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τώρα θα ακούσουμε κάποιους αγορητές. Συνάδελφε Κοκ, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, όταν πριν από 25 χρόνια ξεκίνησα τη θητεία μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα άτομα με αναπηρίες ή με ειδικέ ανάγκε δεν μα απασχολούσαν. Ήταν αόρατοι οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτό οφειλόταν και στο γεγονό ότι δεν υπήρχε καμία επιδίωξη οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα. Αυτό το φράγμα το έχουμε ξεπεράσει. Το 2020 θα έχουμε στην Ευρώπη 120 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες όλων των ε, επιπέδων και όλων των κατηγοριών. Άρα η έκθεση αυτή μας αφορά όλους και όχι μόνο τα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Στις ε, μεταφορές, ε, στις θαλάσσιες, οδικές και ναέρες μεταφορές υπάρχουν ήδη κανόνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα. Οι νέοι κανόνες λοιπόν συμπληρώνουν αυτούς τους ήδη υπάρχοντες κανόνες και αυτό το χαιρετίζω. Ήταν αναγκαίες αυτές οι συμπληρώσεις όπως για παράδειγμα ε, να συμπεριλαμβάνονται πλέον ε, στις απαιτήσει ε, και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης σε αεροδρόμια και λιμάνια. Ιδίως με χαροποιεί το γεγονός ότι η στρατηγική αυτή συμπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα όλων των ανθρώπων να χρησιμοποιούν τον αριθμό έκτακτη ανάγκη 112. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί μια αυτόνομη ζωή για όλα τα άτομα με αναπηρίε. Και νομίζω ότι θα αποτελέσει η πράξη αυτή τη βάση επί τη οποία θα εργαστούμε στα ε, τα επόμενα χρόνια. Και το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση της σημασίας αυτών που λέω. Ευχαριστώ συνάδελφε Ντάντη για ένα λεπτό Νικόλα, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητα θα δώσει απτά θετικά αποτελέσματα για πάνω από 80 εκατομμύρια ανθρώπου που στην Ευρώπη πλήττονται από κάποια αναπηρία ή ε, κάποια κινητικό περιορισμό. Υπολογιστέ, κινητά και τραπεζικέ υπηρεσίε τερματικά αυτοεξυπηρέτηση θα πρέπει να σέβονται τι προποθέσει αυτέ για προσβασιμότητα που θα είναι εναρμονισμένε οι απαιτήσει για να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη στο shopping, στο διαδίκτυο, μεταφορές, ε, ε, τραπεζικές υπηρεσίες, ενιαίο αριθμό ανάγκης όλοι οι πολίτες ακόμα πιο ευάλωτοι θα μπορούν να έχουν τις ίδιες συνθήκες ε, προσβασιμότητας στην ίδια τιμή. σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο όσον αφορά το χρόνο εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών που είναι πολύ μακρά διαρκείας και όσον αφορά τι προαπαιτήσει για, την, για το περιβάλλον, για τα κτίρια, προσβασιμότητα στα κτίρια. Εκεί το Κοινοβούλιο είχε προτείνει κάτι καλύτερο από αυτό που βγήκε από τον τριμερή διάλογο. Όμω η οδηγία για την προσβασιμότητα, παρόλο που δεν είναι επαρκή, επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη είναι πιο δίκαιη σε επίπεδο ανθρώπου και εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν περισσότερη ανάγκη. Ευχαριστώ κύριε Ντάντη. Συνάδελφε Πιετικάνιν, έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Κυρία Πιετικάνιν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Δέκα χρόνια παιδευτήκαμε με τις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες και επιτέλους μπορούμε να το στηρίξουμε. Αυτό όμω αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους πιο φυσιολογικά, τα κτίρια, ε, τα σπίτια, τα προϊόντα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Γιατί οι ψηφιακές υπηρεσίες ε, δυστυχώς αποκλείουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι τεχνολογίες ε, των πληροφοριών μπορούν να βοηθήσουν και τα άτομα με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Αλλιώς υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους, αποκλείονται. Το επόμενο βήμα λοιπόν, σε επίπεδο χωρών μελών, πρέπει να γίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να λάβει υπόψη τις ανάγκες αυτών των ομάδων ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένους κλπ. Χρειάζεται να αναπτύξουμε τα κατάλληλα προϊόντα και τις υπηρεσίες ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Στέγαση επίσης είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα που να αποκλεί ε, τα άτομα ε, με αναπηρίες είτε δεν βλέπουν αρκετά, είτε έχουν πρόβλημα ακοής, να φροντίσουμε να μπορούν όλοι να έχουν εξίσου πρόσβαση. Τώρα πάμε στη δικασία Catch the Eye. Συνάδελφε Στίβενς, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη έχουμε 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες και 150 εκατομμύρια ηλικιωμένου. Κάθε νομοθεσία λοιπόν που φροντίζει για πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες για αυτούς είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Χαίρομαι λοιπόν που αυτό το θέμα προχωράει όσον αφορά την προσβασιμότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πάει αρκετά μακριά κατά τη γνώμη μου. Αν συγκρίνουμε με το τι γίνεται στις ΗΠΑ, η Ευρώπη βρίσκεται πολύ πίσω όσον αφορά την πλήρη προσβασιμότητα. Στι ΗΠΑ υπάρχει η πράξη για τους Αμερικανούς με αναπηρία που αποτελεί μια νοοτροπία πλέον. Και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τις ιδιωτικέ επιχειρήσεις και όλους που είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ευκαιρίες και προσβασιμότητα. Η νοοτροπία αυτή είναι που λείπει εδώ. Και έτσι τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια. Δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Είναι πραγματικά κρίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στίβενς. Συνάδελφε έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πράγματι, πρέπει να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα για τα άτομα ε, με αναπηρίες κυρίως. Αλλά βέβαια να ρωτιέμαι, μήπως, μήπως μια νομοθεσία όχι από πάνω προς τα κάτω θα βοηθούσε. Αν ε, οι παράγοντες του εμπορίου, επιχειρήσεις που είναι πιο κοντά στους ε, καταναλωτές, ε, θα ήταν αυτοί που θα έπρεπε να φροντίσουν για αυτή την προσβασιμότητα και όχι από πάνω προς τα κάτω. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε με αυτό τον τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ε, την κίνηση του νερού. Αντί να καθόμαστε να τα σκεφτόμαστε έτσι για το μέλλον, πώς θα έπρεπε να φροντίσουμε να προσφέρουμε περισσότερη ευελιξία στις επιχειρήσεις γιατί αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε από πάνω προς τα κάτω. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό παρακαλώ. Grazie, Presidente. Πράγματι, όπως υπόθηκε, υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς, και άλλα 150 εκατομμύρια οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι. Και είναι δεδομένο ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για να υπάρξει πλήρης προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι τα ΑΜΕΑ πραγματικά έχουν δυσκολίες για να συμμετάσχουν στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή της ευρωπαϊκής ένωσης και γι' αυτό απαιτούνται πολύ συγκεκριμένα μέτρα. και έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες κύριε πρόεδρε τις οποίες έχουμε λάβει στην επιτροπή αναφορών από χιλιάδες πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης. νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει η εξή ρύθμιση να μην χρηματοδοτείται κανένα έργο είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό με κοινοτικού πόρους με πόρους της ευρωπαϊκής ένωσης εάν δεν υπάρχει η ρύθμιση για πλήρη προσβασιμότητα. αυτό πρέπει να είναι κριτήριο προκειμένου να εγκριθούν οι διάφορες χρηματοδοτήσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Λόκεγκαρτ για την ε, θέση του, τη τόσο επικοδομητική και παρά το Συμβούλιο κατάφερε να πετύχει την καλύτερη δυνατόν συμφωνία. Πρόκειται για την αναγνώριση των τόσων εκατομμυρίων Ευρωπαίων που υποφέρουν από κάποιο βαθμό αναπηρίας. Και έτσι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο τρόπο θα ισχύουν υποχρεώσει που έχουμε βάσει του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίε. Είτε πρόκειται για τι μεταφορέ, είτε πρόκειται για βασικές υπηρεσίε, ψηφιακέ ή όχι. Ακόμα και στου υπολογιστέ, τα τερματικά, τα τηλέφωνα ή τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ένα άλλο μεγάλο επίτευγμα είναι ότι είναι προσβάσιμες οι υπηρεσίες του 112. Κρίμα που δεν συμπεριλαμβάνονται τουριστικές υπηρεσίες, τις παραλίες για παράδειγμα ή άλλου είδους ψυχαγωγία. Είναι ένα καλό βήμα. Μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη θέση παγκοσμίω χρησιμοποιώντας τεχνολογίες οι οποίες βοηθούν τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ, ήταν τελευταία παρέμβαση και τώρα ο Επίτροπος ο κ. Μίμητσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές, έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ήταν εντατικές. Χρειάστηκε όλοι να δείξουμε ευελιξία και προθυμία για να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί από εσά θα, είχα, θα προτιμούσατε να καλύπτονται από τη νομική αυτή πράξη περισσότεροι τομεί ή να υπήρχε περισσότερη φιλοδοξία σε κάποια ζητήματα. Πραγματικά, η πρόταση της Κομισιόν ήταν πιο φιλόδοξη. Οπότε συμμερίζομαι και κατανοώ κάποιες από τις ανησυχίες σας. Όμως το τέλειο μερικές φορές είναι ο αντίπαλος, ο εχθρός του καλού. Και πρέπει τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε την σημαντική προόδο που έχουμε σημειώσει και που θα σημειώσουμε. Η προσβασιμότητα πολλών προϊόντων και υπηρεσιών στην καθημερινότητα θα ωφελήσει όλους τους πολίτες. Όλοι πρέπει να ωφεληθούν από την ψηφιακή επανάσταση. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω, καθώς οι κοινωνίες μας αλλάζουν. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, οι αλλαγές αυτές όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας είναι προφανείς, προφανώς θετικές και προφανώς αναγκαίες. Είναι τόσο αναγκαίες και θετικές που οι πολίτες σε λίγο καιρό θα αναρωτιούνται γιατί δεν είχαμε αυτές τις απαιτήσει και νωρίτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο και τώρα στον εισηγητή θα δώσουμε το λόγο. Ο κ. Λόκεργαντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην συζήτηση την οποία παρακολούθησα με προσοχή. Οι διαπραγματεύσεις, όπως υπόθηκε, συνεχίστηκαν για πάρα πολλά χρόνια. Το ποτήρι είναι πάντοτε μισοάδιο ή μισογεμάτο. Εγώ ανήκω σε εκείνους που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Όπως και ο Πίτροπος Μίμητσα, θεωρώ ότι έχουμε καταλήξει σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και ίσως το καλό είναι, όπως είπατε κι εσείς, ε, το τέλειο μάλλον είναι ο εχθρός του καλού. Βρισκόμαστε σε κάθε περίπτωση σε μια κατάσταση όπου έχουμε ξεπεράσει πλέον την στασιμότητα που μας χαρακτήριζε για δεκαετίες. Πριν από 20 χρόνια δεν ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε τη θέση στα άτομα που, με αναπηρία που τους αξίζει. Μπορούμε τουλάχιστον σήμερα να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε διανύσει αυτό το δρόμο, ότι έχουμε πλέον φτάσει σε αυτό το σημείο όπου μπορούμε πια να προσφέρουμε αξιοπρεπείς όρους καθημερινής διαβίωσης σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους και την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ξέρω ότι πολλοί θα θέλαμε να είχαμε επιτύχει περισσότερα και εγώ ε, θα ήθελα να είχαμε επιτύχει περισσότερα. Όμως νομίζω ότι μπορούμε τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος τέθηκαν αυτά τα ζητήματα, συζητήθηκαν επί μακρόν και φαίνεται ότι και στα κράτη-μέλη έχει ξεκινήσει μια αντίστοιχη συζήτηση. Θεωρώ ότι η νομική πράξη αυτή θα τύχει ευρεία υποστήριξη. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που έκανε. Πέρα τούτη η συζήτηση, ευχαριστώ τον Επίτροπο τον κύριο Μίμητσα, ο οποίο ε, ήρθε μαζί μα σήμερα το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε ε, τη δήλωση της, ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επίγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητε. Χαιρετίζω την Επίτροπο κυρία Γιούροβα που ήρθε εδώ και δίνω το λόγο εν ονόματι του Συμβουλίου στον Υπουργό, στον Τσότ. Έχετε το λόγο, κυρία Υπουργέ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον πρόεδρο Ταγιάννη για την επιστολή του. Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Να βρω το σωστό χαρτί, παρακαλώ. Sorry, Okay, sorry for this. Συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ που καλέσατε την Προεδρία να έρθει να συνεισφέρει στη συζήτηση αυτή και θα αρχίσω αναφέροντα ρητά ότι το Συμβούλιο έχει δεσμευθεί στην καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Η Προεδρία και το Συμβούλιο ολόκληρο συμμερίζονται το επίγον του ζητήματος και χαίρεται για τη δέσμευση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταπολεμήσουν την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Έτσι λοιπόν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή συνεργάζονται όλα αυτά τα χρόνια για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. Να έχουμε δηλαδή ένα καθεστώς που θα καταπολεμά την νομοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το 2019 εγκρίνουμε τις τελευταίες τροπολογίες στην οδηγία για την καταπολέμηση του νομοποίησης σε παράνομου χρήματος που αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της καλής συνεργασίας. Βέβαια χρειάζεται περισσότερη πρόοδος στην καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Ποια είναι τα ζητήματα. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με την κατεξοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρίτες ε, χώρες. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει βέβαια ότι ο κατάλογος δεν αποτελεί βασικό στοιχείο του έργου μας. Αντίθετα, αλλά για να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Και ακριβώς αυτό είναι που αναφέραμε και εμείς στη δήλωσή μας στο Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι προκειμένου να έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό προτείνεται με διαφανή τρόπο να προχωρήσουμε και με τρόπο όπου θα δώσουμε την ευκαιρία και στις διάφορες χώρες να αναλάβουν δράση. Γι' αυτό και το Συμβούλιο ζητάει ένα νέο κατάλογο, μια νέα ενωσιακή λίστα, η οποία θα ενισχύει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είμαστε ενωμένοι και έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε την συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Προχωρούμε και σε άλλα μέτωπα επίσης για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Και ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσει αυτέ τι μέρε για ένα σημαντικό, μια σημαντική νομοθετική πράξη για την καταπολέμηση νομοποίηση παράνομου χρήματος. Οι χώρες μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρουν και δίνουν πολύ μεγάλη ε, σημασία σε αυτό το φάκελο. Εξάλλου το Συμβούλιο αποφάσισε το Δεκέμβριο να αφιερώσει πολλή προσπάθεια στην καταπολέμηση αυτή προκειμένου να βελτιωθεί το τρέχον σύστημα και ελέγχουμε τις εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, προσβλέπω στις δικές σας απόψεις και στις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχιση της συνεργασίας μας για την νέα αυτή ενωσιακή λίστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα στην ε, ημερήσια διάταξή μας είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής το επίγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, το λόγο έχει η κυρία Τσιώτη. Συγγνώμη, το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής η Επίτροπος Βέρα Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ που οργανώσατε την σημερινή συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για το γεγονός ότι συμμερίζεται τον επίγοντα χαρακτήρα του θέματος. Μετά από κάθε τρομοκρατική επίθεση ακούμε παθιασμένες ομιλίες για το πώς πρέπει αποτελεσματικά να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες. Έπειτα από κάθε τραπεζικό σκάνδαλο ακούμε ε, ομιλίες, πύρινες για το ότι πρέπει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να γίνει πιο υγιής. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μέσω των ε, καταλόγων τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου. Και αυτό κάναμε βάσει μιας μεθοδολογίας η οποία υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε με κάθε διαφάνεια. Γι' αυτό και ξεκινώ ε, εκφράζοντας την ε, δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι ο κατάλογος αυτός ε, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο, διότι το να είχαμε ένα τέτοιο κατάλογο θα μας ε, επέτρεπε άμεσα να ξεκινήσουμε αποτελεσματικά ε, τον αγώνα αυτών. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά έχουμε θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά μας την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και της, του ξεπλήματος χρήματος. Και πάντοτε είχαμε την πλήρη υποστήριξη και των ευρωβουλευτών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μια σειρά από τρομοκρατικές υποθέσεις στην Ευρώπη και είδαμε μεγάλα σκάνδαλα ξεπλήματος χρήματος ε, για το πώς ε, το οργανωμένο έγκλημα καταχράτε το οικονομικό, σας, το οικονομικό μας σύστημα. Δουλέψαμε ακούραστα για να καταστήσουμε το σύστημά μας πιο ανθεκτικό ε, και για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Δύο φορές επικαιροποιήσαμε την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Και έχουμε προσωρινά έρθει σε συμφωνία για μια νέα οδηγία για την χρήση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών από τις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτή τη, δε, ε, αυτή τη βδομάδα δε βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής που, αρχής που θα ε, δώσει μεγαλύτερο ρόλο στην ε, εποπτεία του χρηματοπιστικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της, του ξεπλήματος χρήματος. Η, ο κατεξοδότηση κανονισμός που ενέκρινε η Επιτροπή στις 20 Φεβρουαρίου ε, που περιλαμβάνει την, ε, τις χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα αποτελούν, ε, αποτελεί μία από τις προσπάθειες για την προστασία του Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από τις απειλές της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του ξεπλήματος χρήματος. Δυστυχώς όμως η πράξη αυτή δεν θα τεθεί σε ισχύ για τους λόγους που ανέφερα ε, αρχικά. Το Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου εξέφρασε την αντίρρησή του ως προς την έγκριση αυτού του κατεξιδότηση κανονισμού. Δυστυχώς, όπως είπα, είμαι πολύ απογοητευμένη από αυτή τη στάση του Συμβουλίου και, το ζήτημα, και για το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο ούτε από τους Υπουργούς Οικειοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε και στο ΕΚΟΦΗΝ που έγινε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στην ε, πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είχαν συναποφασίσει να αυστηρίνουν τους ε, κανόνες μέσω και της δημιουργίας μιας σχετικής task force. Εμείς θέλουμε ε, να υπάρχει πολυμέρεια και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η δουλειά της Task Force, της οποίας αποτελούμε ιδρυτικό μέλος και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα των εργασιών της. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα βήματα για να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης ε, όπως ακριβώς ε, περιλαμβάνονται στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης ε, παράνομων εισόδων. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από το σκάνδαλο των Panama Papers, εμείς και εσείς είχαμε ε, συναποφασίσει να θεσπίσουμε κανόνες διαφάνειας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάτι που βεβαίως υπερβαίνει τους κανόνες της Task Force. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλώς να ε, αναπαράγουμε τη λίστα της Task Force. Έχουμε νομική υποχρέωση να προβούμε σε δική μας αυτόνομη αξιολόγηση και για να ξεκινήσουμε, για να καταρτήσουμε αυτόν τον νέο, τον πρώτο κατάλογο η Κομισιόν βάσει ε, μιας, πολύ, μιας πολύ ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ε, ε, προχώρησε στην, στο έργο αυτό, πάντοτε σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τους. Η Κομισιόν επίσης ήρθε σε επαφή και με τρίτες χώρες που εμπλέκονται αμέσως αφότου το Σώμα των Επιτρόπων κατέληξε στην προσωρινή λίστα στις 23 Ιανουαρίου σεβόμενο το δικαίωμα των τρίτων χωρών να ακουστούν οι δικές τους θέσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με τις χώρες που αφορά η, η, λίστα αυτή, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα και θα, τις, ε, θα συνεχίσουμε να τις βοηθούμε για να άρουν τα προβλήματά τους. Δεν βάζουμε χώρες σε τέτοιους καταλόγους απλώς και μόνο για να το κάνουμε, αλλά για να προστατεύσουμε το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ω επόμενα βήματα, σε πολιτικό επίπεδο, θα έρθουμε στη συζήτηση με εσά και με το Συμβούλιο για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Στόχο μα είναι να ανταποκριθούμε πλήρω στι νομικέ μα υποχρεώσει που απορρέουν από την οδηγία. Είναι κοινή μα υποχρέωση ω θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε του πολίτε και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των απειλών τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και τη διαφθορά. Ταυτόχρονα σας ζητώ να μου δώσετε την ευκαιρία να οριστικοποιήσουμε τον κατάλογο αυτό εντός της θητείας. Γιατί θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου και το τραπέζι των εργασιών μας εντός αυτής της θητείας. Και επαναλαμβάνω ότι για να επιτύχω αυτόν τον στόχο χρειάζομαι οπωσδήποτε την υποστήριξή σας. Προτιμα... Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει ο κύριος Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η καταπολέμηση του μαύρου χρήματος χρειάζεται, χρειαζόμαστε μια, μια λίστα τρίτων χωρών η οποία θα είναι αξιόπιστη. Και ακριβώς επειδή είχαμε στο παρελθόν και ε, εμείς τις αντιρρήσεις μας για προηγούμενες εκδοχές αυτή τη λίστα, είχαμε και εμείς αναπέμψει ε, στην Κομισιόν τέτοιες προσωρινές λίστες Είχαμε πει δε τότε ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουμε copy-paste τις λίστες της Task Force. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόνομα να καταρτήσει τη δική της λίστα τρίτων χωρών. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Γιατί δεν υπάρχουν στη λίστα αυτή χώρες όπως η Ρωσία. Επίσης υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα, Πώ μπορεί κανείς να ενταχθεί ή να αφαιρεθεί από τη λίστα. Όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν. Ταυτόχρονα ομω έχω ε, την αίσθηση ότι η απόρριψη τη του, της λίστας αυτής από το Συμβούλιο ήταν κάπως αδιαφανής. Ε, και τις τελευταίες εβδομάδες πολλές φορές το επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν να μπει μία ή άλλη χώρα σε αυτή τη λίστα γιατί είναι σημαντική εταίρη μας. Ναι, αν ακολουθήσουμε όμως αυτή την επιχειρηματολογία, η αξιοπιστία της λίστας αυτής μπορούμε να την πετάξουμε στα σκουπίδια. Γιατί είναι σαφές ότι χρειάζεται απλώς να κάνει κάποιος, κάποια χώρα δουλειά λόμπι για να αφαιρεθεί από τη λίστα. Δεν μπορεί αυτός να είναι ο στόχος, διότι σε τελική ανάλυση στόχος μας είναι ε, να εξασφαλίσουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνεται αντικείμενο κατάχρηση για τη χρηματοδότηση της ή για την διαφθορά. Δεν αρκεί ε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να έχει νέες αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της, ε, του ξεπλήματος χρήματος και ταυτόχρονα να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για την κατάρτιση μιας λίστας τρίτων χωρών. Καλό την Επιτροπή να υποβάλει ταχύτατα τη νέα της πρόταση και το Συμβούλιο να συμφωνήσει. Κρατών το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν στρατηγικά προβλήματα όσον αφορά το μέτρο αυτό. Βάσει ανεξάρτητων αξιολογήσεων, έχουμε την οδηγία για την ε, αντιμετώπιση πολέμηση της νομοποίησης ε, εσόδων που σίγου, από παράνομες δραστηριότητε που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι πολύ σημαντική και η φοροδιαφυγή προς ε, φορολογικούς παραδείσους. Για άλλη μια φορά, οι προσπάθειες για διαφάνεια, για φορολογική δικαιοσύνη μπλοκάρονται από τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο. Πρόκειται για συλλογική ευθύνη. Μην έρχονται λοιπόν στις Βρυξέλλες μετά και να μας λένε ότι φταίνει οι Βρυξέλλες. Δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τον λαϊκισμό με αυτόν τον τρόπο. Το Συμβούλιο φταίει. Όλες καθεμία χωριστά και όλες οι κυβερνήσεις των χωρών μελών που συμπεριφέρονται φιλικά απέναντι σε κυβερνήσεις όπως είναι της Σαουδικής Αραβίας ή απέναντι στο Τραμπ. Κυρία Επίτροπε, χαίρομαι για την αποφασιστικότητά σας και την επιμονή σας. Να ξέρετε ότι μας έχετε μαζί σας. Την ομάδα των συντηρητικών, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχεται η Ευρώπη τώρα με ένα νέο κατάλογο, μια νέα ενωσιακή μαύρη λίστα. Ωραία. Κάναμε καλά τη δουλειά μας. Πάντα μπορούμε να την κάνουμε καλύτερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως αυτές τις ε, δύο εβδομάδες καθόρισε ένα τέτοιο κατάλογο χωρίς ε, μεθοδολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι τα έχει καταφέρει καλύτερα. Υπάρχει ένας νέος κατάλογος, ο Παναμά κλπ. Προβλέπονται κυρώσεις, αλλά οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να εμφανίζουν τις συναλλαγές, να τις ελέγχουν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταπολεμηθεί η οικονομική απάτη. Το κόμμα μου έχει δεσμευτεί σε αυτόν τον αγώνα εδώ και χρόνια. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Τόλβας για δύο λεπτά. Λοιπόν, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διάβασα τον κατάλογο αυτό. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Και γιατί? Διότι εδώ και αρκετό καιρό συζητάμε, εδώ με τη συνάδελφο, εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να συζητάμε. Πάνε έξι χρόνια τουλάχιστον. Υπήρχαν διάφοροι κατάλογοι, δεν είχαμε καταφέρει να οργανωθούμε. Τώρα όταν κοιτάζω τον κατάλογο αυτό, αναρωτιέμαι γιατί διαλέγουμε κάποιες χώρες και δεν διαλέγουμε κάποιες άλλες. Εκπλήσωμα ακόμα περισσότερο. Γιατί ε, διαπιστώνουμε ότι έχουν υπάρξει ένα σωρό οικονομικά σκάνδαλα που βασίζονται στο ίδιο πάντα μοντέλο. Πρόκειται για τη Ρωσία. Ίσως αυτοί οι οποίοι συνέταξαν τον κατάλογο να μην γνωρίζουν πολύ καλά το ρωσικό σύστημα. Εγώ όμως έχω περάσει έξι χρόνια και με εκπλήσει ειλικρινά που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ακόμα πιο σοβαρά αυτό το πρόβλημα. Γιατί πάντα υπάρχει ένα οργανωμένο έγκλημα από τη Ρωσία. Κλέβονται χρήματα και τελικά αν κοιτάξετε καλά θα δείτε ότι πάντα υπάρχει το ίδιο νήμα που οδηγεί εκεί σε κάθε οικονομικό σκάνδαλο. Οπότε με εκπλήσει που δεν βλέπω τη Ρωσία σε αυτό το κατάλογο. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πραγματικά σοβαρά δεν το έχετε λάβει υπόψη σας. Μα τα χρήματα πάντα επιστρέφουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία και γι' αυτό δεν μας εμπιστεύεται πια ο κόσμος. Πρέπει να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν δράσουμε ε, διεθνώς. Οι πολίτες μας πρέπει να καταλάβουν, έτσι θα μας εμπιστευτούν, αν πιστέψουν ότι πραγματικά καταπολεμούμε την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολεμούμε και τους φορολογικούς παραδείσους. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Γκίγκολτ. Κύριε Πρόεδρε, αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες ε, είναι πραγματικά ε, απίστευτα. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στο Συμβούλιο. Έχουμε καταλήξει από κοινού σε μεθοδολογία. Η Κομισιόν ε, ε, ξεκίνησε το έργο της. Για μήνες δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Όταν άρχισε λίγο-λίγο να γίνεται γνωστή η, λύση, η λίστα, άρχισαν να υπάρχουν παρεμβάσεις από τον Παναμά, από κτίσεις των ΙΠΑ και από τη Σαουδική Αραβία. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια κριτική επί της μεθοδολογίας, η οποία είναι τελείως αναξιόπιστη. Διότι μέχρι σήμερα Καμία από τις αξιολογήσεις της Κομισιόν για τις επιμέρους χώρες δεν έχει ε, δεχθεί συγκεκριμένη αντικειμενική κριτική. Αντιθέτως, απλά απορρίπτει το Συμβούλιο τη λίστα ε, αυτή των, των τρίτων χωρών. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι. Το είπε και η Κομισιόν για την ε, Ρωσία, για τα Εμμυράτα, για το Αιζερβαϊτζάν. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αξιολόγηση. Δεν είναι δυνατόν τώρα να σταματήσουμε. Πρέπει αντιθέτως να συνεχιστεί το έργο αυτό, να καταλήξουμε μία, μία λίστα χωρών και η Κομισιόν πρέπει επιτέλους να δημοσιοποιήσει ε, αυτόν τον κατάλογο των χωρών, των τρίτων χωρών. Ε, Ευρωπαϊκής Αριστεράς, το λόγο έχει ο κύριος Κάρθη για ένα λεπτό. Έχουμε μπροστά μας ένα από τα πιο μεγάλα αποτελέσματα ε, όσον αφορά τις πιέσεις των λόμπι στο, στο Συμβούλιο που είναι βλαβερά για το λαό της Ευρώπης. Η νέα μαύρη λίστα δεν είναι τέλεια πρόταση. Αγνοεί το γεγονό ότι η πλειοψηφία των σκανδάλων για το ξέπλυμα χρήματο τα πρόσφατα χρόνια ενέπλεκαν ευρωπαϊκέ τράπεζε. Παρ' όλα αυτά, ευπρόσδεκτη η αύξηση τη αυτονομία στη διαδικασία, οι στόχοι του αντιρρήσει του Συμβουλίου έχουν πολιτικά κίνητρα, είναι παρεμβάσει σε μια διαδικασία που υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη. Ιδιαίτερα ανησυχώ διότι ε, η προάσπιση τη Σαουδική Αραβία και των ΗΠΑ από ευρωπαϊκέ κυβερνήσει είναι αποτέλεσμα των δεσμών του των εμπορικών και των τραπεζικών και των λόμπι των Αμερικανών και τη Σαουδική Αραβία. Δεν χρειαζόμαστε ένα μαύρο κατάλογο κατεπηγόντω, αλλά χρειαζόμαστε μηχανισμού για να αποφύγουμε το λόμπι που ασκούν οι εταιρείε σε διάφορε χώρε και αυτό είναι επιβλαβέ του δημόσιου συμφέρον και θα πρέπει να έχουμε πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία των λόμπι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας. Το λόγο έχει ο κύριος Κόμπερν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι σοσιαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αιμονή με το ξέπλυμα. Μην και χαθεί έστω και μία δεκάρα από φορολογικά έσοδα. Κάποιοι όμως πάντοτε θα μπορέσουν να φοροαποφεύγουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να το ελαχιστοποιήσουμε το, το φαινόμενο αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και να συνεχίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να σταυρώνουμε τον κάθε τίμιο επιχειρηματία με γραφειοκρατικούς κανόνες που τάχα καταπολεμούν το ξέπλυμα χρήματος. Οι επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης εμείς δεν είμαστε τόσο νευρωτικοί με το ξέπλυμα χρήματο και γι' αυτό και έχουμε χαμηλότερη ανεργία. Έχουμε πολύ μικρότερη ανεργία από την Ιταλία και την Γαλλία. Η εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης γίνεται μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, όχι μέσω της αύξησης. Αυτό ωφελεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Η σοσιαλιστική ζήλια ε, των Ευρωπαίων κατά των ε, επιτυχημένων επιχειρηματιών τελικά στρέφεται κατά των ίδιων των πολιτών. Θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας, να μας καταστήσει ένα κράτος κατασκόπων. Ταυτόχρονα όμως οι τραπεζίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και μετά το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν ε, ασυλία. Αυτή είναι η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει ένας κανόνας για μας και ένας κανόνας για όλους τους υπόλοιπους. Και της ελευθερίας, το λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παριστάμεθα σε ένα θέαμα πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό το παιχνίδι των χωρών είναι ένα σαν παιχνίδι, σαν χαρτοπέγνιο που μπαίνουν οι χώρες και βγαίνουν από τη λίστα και δείχνουν την ελάχιστη βούληση για παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για να τόσο ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Αλλά πρέπει αρκεί να θυμίσουμε το συναγερμό που χτύπησε στις επιτροπές μας από μια προσωπικότητα τον τότε διευθυντή καταπολέμηση των ναρκωτικών στις Γενέβη, στις υπηρεσίες που έλεγε ότι όλο το διεθνές εμπόριο των ναρκωτικών περνά από την ανακύκλωση του τραπεζικού συστήματος, από κάποιους τομείς του χρηματοστατικού και τραπεζικού συστήματος. Όσο διαρκεί αυτή η αδιαφάνεια η δημοσιονομική ε, και έχουμε τα offshore, τις εταιρείες offshore, πώς θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει με σαφή και αποφασιστικά μέτρα και να εφαρμόσει και να ξεφύγει από όλα αυτά τα, τις προδιαγραφές που είναι διάτριτες που έχουν οι χώρες που διευκολύνουν το εμπόριο ναρκωτικών λοιπά μέσω αυτής της αδιαφάνειας και του ξεπλήματος χρήματος. Θα ήθελα να πω στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ευγενέστατη κυρία, ότι η πέμπτη οδηγία θεσπίζει σαν ποιοτικό στοιχείο το, το, το, τη εταιρεία, την πραγματική ιδιοκτησία. Και κλείνω. Κλείνω. così agevole risalire i veri proprietari delle società offshore. È così sicura che nei nostri paesi sia possibile, i paesi dell'Unione Europea, prima di andare a cercare i Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Σας παρακαλώ όλους να τηρείτε το χρόνο γιατί δεν έχουμε περιθώριο χρόνου είμαστε λίγο εκτός χρονοδιαγράμματος. Προχωρούμε με τον κύριο Ρωσάτη για 1,5 λεπτό. Thank you. Uh, thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Γιούροβα για το γεγονός ότι δίνει στους Ευρωπαίους πολίτες αυτό που ζητάμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έναν πραγματικό ευρωπαϊκό ε, κατάλογο χωρών που εμπλέκονται στο ξέπλυμα χρήματος. Και αυτό βάσει της αξιολόγησης που διενήργησε η Κομισιόν για τις διάφορες χώρες. Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, κυρία Γιούροβα. Ταυτόχρονα θέλω να πω στους συναδέλφους ότι με την ομάδα μου δυστυχώς ε, ε, είμαστε πολύ ε, απογοητευμένοι που, απε, που απερίφθη από το Συμβούλιο η λίστα αυτή, γιατί αυτός ο μαύρος κατάλογος, ο, ο προσδιορισμός μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών θα ήταν πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι λοιπόν ένα εμπόδιο που μας βάζει εδώ σε αυτόν τον δρόμο το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι ε, χαιρετίζω την έως σήμερα μεθοδολογία, θέλω να καλέσω την Κομισιόν να λάβει υπόψη τη τα διδάγματα και τα πορίσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή του Κοινοβουλίου Τάξε 3. Να σα υπενθυμίσω ότι όλα τα σκάνδαλα που είχαμε σε αυτή τη θητεία χρηματοπιστωτικά είχαν σχέση είτε με τη Ρωσία είτε με, είτε με Ρώσους πολίτες, με ρωσικά κεφάλαια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν απαιτούν και περιμένουν να δραστηριοποιηθείτε με ε, θάρρος, σε αυτό, τον, αυτό το αντικείμενο και να υποβάλλετε γρήγορα μια καινούρια πρόταση. για λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Γιούροβα, στη θητεία αυτή πολλές φορές εκφράσαμε την δυσαρέστησή μας επειδή δεν υπάρχουν αποτελέσματα και επειδή το Συμβούλιο μπλοκάρει την κατάσταση. Όμω, ο απολογισμός τελικά όσον αφορά τα αποτελέσματα από την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και χρηματοδότησης τρομοκρατίας ε, είναι κάτι σημαντικό. Έχουμε την πέμπτη τέτοια οδηγία η οποία αρχίζει να αποφέρει καρπούς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οδηγία για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, που είναι και αυτός ένας μηχανισμός πάρα πολύ σημαντικός για να προσεγγίσουμε την ε, νομοθεσία, την ποινική των χωρών μελών. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνεισφέρει. Η Σοσιαλιστική Ομάδα έχει στηρίξει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες με μεγάλη επιμονή και με τις επιτροπές τα ξένα 2 και τρία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πρέπει να συνεχίσει να πιέζει το Συμβούλιο έτσι ώστε να μην προσπαθεί να μειώνει αυτόν τον κατάλογο που με αυτόν τον τρόπο δεν καταπολεμάμε το φαινόμενο, αντίθετα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να θεωρηθεί ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική. 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχαμε στην Ισπανία τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση με πάρα πολλά θύματα. Να το θυμόμαστε και αυτό. Το λόγο έχει η κυρία Σαρτσεντίν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλάει όλες τις γλώσσες η κυρία Σούιτς ή δεν ακούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μετά περιμένω ότι θα μας ακούσετε και θα μας ε, απαντήσετε. Γιατί εσείς τα βάζετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τηρεί την ε, νομοθεσία. Εγώ ήμουν εισηγήτρια την προηγούμενη φορά που είχαμε προσπαθήσει με την οδηγία για να καταπολεμήσουμε το κλιματικό χρήμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο όμως δεν πηγαίνει αρκετά γρήγορα και το έχουμε καταδείξει ξανά και ξανά και με το Τσάρλι Εμπδό και με το Μπατακλάν. Μετά από αυτές τις επιθέσεις, εμείς επιμείναμε ξανά και ξανά. Η Επιτροπή κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Και εμείς θέλουμε να καταπολεμηθεί η νομοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα. Αλλά το Συμβούλιο ε, δεν προχωράει. Οπότε, να μας ε, εξηγήσετε ποιο είναι το πρόβλημα της Σαουδική Αραβία, τον Παναμά, και τα διάφορα νησιά, γιατί δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Λόγο έχει ο κύριος Σούρμπαν Κρέσπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια αυτής της